Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μλίναρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και τώρα θέλω να απευθύνω ένα έπαινο σαφέστατο προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγγελα Μέρκελ, διότι δεν έχει οξύνει την προσφυγική κρίση, ούτε έχει προσκαλέσει τον κόσμο όλο στην Ευρώπη, όπως συχνά κατακρίνεται γι' αυτό. Απλώς έδωσε μια Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτό θα πρέπει όλοι οι κυβερνώντες να το σημειώσουν, ότι δικαίωμα στο άσυλο είναι ουσιαστικό ε, συστατικό του καταλόγου αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει μια λύση σε συνεργασία με την Τουρκία. Είναι και αξίζει να υποστηριχθεί και χαίρομαι που αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εδώ με την κυρία Μέρκελ και να ακούσουμε τα σχέδιά της για τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα χαίρομαι που θα έρθει και ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά ε, Ολόντ του οποίου βέβαια τι δραστηριότητε, εγώ τις βρίσκω λιγότερο αξιέπαινε. Πριν από 15 μέρες πήγα στο Καλέ και πρέπει να πω ότι είναι πονίδιστε και πέσχυντες στι συνθήκε για ευρωπαϊκό κράτο που επικρατούν εκεί. Και ε, πριν αρχίσουμε να επικρίνουμε άλλες χώρες να δούμε τα του οίκου μας πρώτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεγιέχικ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να συγχαρούμε και να είμαστε παραστάτες ε, στα κράτη, ε, τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, σωματεία, εργαζομένους και πολίτες ε, που βοηθούν τους πρόσφυγες. Καθήκον της Ένωσης είναι να τους υποστηρίζει και να δίνει τα απαραίτητα κονδύλια που βοηθούν τους πρόσφυγες να ζουν, να στεγάζονται, να εκπαιδεύονται, να μορφώνονται και να βρίσκουν δουλειά. Τα απαραίτητα κονδύλια θα πρέπει ε, να ε, βοηθήσουν για να ξαναδούμε τη λιτότητα που έχουμε επιβάλει σε κράτη, περιφέρειες και ε, οργανώσεις. Χρειάζονται διεθνή προστασία αυτοί οι άνθρωποι που τους έχει βγάλει στο δρόμο ο πόλεμος. Χρειάζεται ασφαλής διάβαση και όχι να αφήνουμε άπλιστους διακινητές να βγάζουν λεφτά στην πλάτη της ένδυας και της απόγνωσης. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων δεν κατακλείζεται ούτε κυριεύεται από 750.000 ακόμα και αν τους υποδεχόμαστε. Όλη η ανθρώπινη ιστορία δείχνει ότι η μετανάστευση δεν είναι βάρος αλλά πλούτος από πλευράς ανθρώπινης, οικονομικής και πολιτισμικής. Η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκπλήσω με πάρα πολύ. Γι' αυτό που ακούω εδώ πέρα για την Ουγγαρία. Υφίσταται επιθέσεις η Ουγγαρία, κατηγορίες με αναλήθειες και ψεύδι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να επικεντρωθούμε στο εξής να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους πρόσφυγες, να τους βοηθήσουμε ε, στους καταβλισμούς εκεί στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι οι πραγματική πρόσφυγες, εκεί που είναι στους καταβλισμούς και όχι αυτοί που έχουν έρθει στα σύνορα και ε, πετροβολούν τους αστυνομικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα τρίτα κράτη εκείνα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανθρωπιστικές ανάγκες και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν εκεί στους καταβλισμούς, δεν ρισκάνουν τη ζωή τους. Δεν ε, κινδυνεύουν. Έτσι μόνο θα αποτρέψουμε ε, όλα αυτά τα δεινά για τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Οι οποίοι καταταλαιπωρούνται, έρχονται εδώ και διαπιστώνουν ότι πρέπει να απελαθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προστατεύουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και καλούμε όλους να το πράξουν. Να τηρούμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να πούμε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τους πάντες. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, κυρία Ζήπελ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων. Και αρχίζω από τις χώρες τη Βαλκανικής. Αν τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε κάνει αρκετά για τον εκδημοκρατισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Βαλκανικής, το κάναμε ή μήπως αδιαφορήσαμε. Ε, Λίβανος, η Ορδανία, είναι μια κατάσταση αφόρητη αυτή που ζουν. Τα παιδιά δεν μορφώνονται. Δεν υπάρχουν επαρκή τρόφιμα και μεταξύ άλλων διότι τα δικά μας κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει ε, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Και οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία δεν μπορούν να ζητήσουν άσυλο, δεν επιτρέπεται να εργάζονται, δεν παίρνουν καμία κοινωνική υποστήριξη και με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούν να παραμείνουν στη σημερινή Τουρκία. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Στη ΔΕΕ... Ευρωπαϊκή Ένωση αποθούνται βία ε, στα σύνορα άνθρωποι, πολλές φορές τους πυροβολούν κιόλα. Η κατάσταση σε Ιταλία και Ελλάδα είναι αφόρητη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολλά κράτη-μέλη για πάρα πολύ καιρό παρέμειναν θεατές όταν δεν ε, ε, έστριβαν τα μάτια προς άλλη κατεύθυνση. Τους έλεγαν, ε, καλά και εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. δείτε εσείς που έχετε εξωτερικά σύνορα πώς θα κανονίσετε την πορεία σας. Τώρα όμως ε, διαπιστώνουμε ότι οι εθνικές απαντήσεις δεν επαρκούν και δεν είναι μόνο η προστασία των ανθρώπων. Ε, αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους είναι η περιχαράκωση των συνόρων μας. Τι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν επιβαρύνεται από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που μέχρι τώρα επιβαρύνεται όμως και δεν έχει καταφέρει να τα βγάλει πέρα είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο που δεν μπορεί να βρει κοινέ ευρωπαϊκές απαντήσεις. Τώρα είναι 12 παρα 5. Τώρα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με κάθε τρόπο, οικονομικά, οργανωτικά, από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ή από πλευράς κρατομελών για την καταγραφή, καταχώρηση, υποδοχή, ε, κατανομή, βοήθεια για τις τρίτες χώρες. Οι πρόσφυγες, οι δικοί μας πολίτες και η Ευρώπη επιτέλους χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι άχρηστη και αναποτελεσματική αυτή η συζήτηση που την έχουμε και επανειλημμένως. Ε, είχαμε πει ότι το Ισλαμικό κράτος ε, θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα τους. Είχαμε μιλήσει για την Τουρκία που βομβαρδίζει Κούρδους στο Ιράκ και ε, λέμε συνέχεια ότι μόνο με στρατιωτική παρέμβαση θα εμποδίσουμε την κρίση και θα σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δυστυχώς όμως τίποτα δεν συνέβη, παρά τις προειδο... τίποτα δεν κάναμε παρά τις προειδοποίησεις. Και η πατρίδα μου, η Βουλγαρία, υποφέρει από τους πρόσφυγες. Ε, δεν υπάρχει κατανόηση. Ε, και δεν γίνεται σωστός διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Οι οικονομικοί μετανάστες προέρχονται από, ασφαλείς, από ασφαλείς χώρες όπως η Τουρκία. Και αφήστε τις ποσοστώσεις και τα hot spot. Μόνο η Γερμανία είναι το hot spot, εκεί θέλουν να πάνε όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σράντο. Η προσφυγική κρίση έχει δείξει την αδυναμία των ευρωπαϊκών μα πολιτικών. Η πολιτική ασύλου δεν είναι καν πολιτική. Είναι ένα πρωτόκολλο που δεν το σέβεται κανένα. Το σύστημα Σέγγεν για τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύθηκε και στα εσωτερικά σύνορα έχει ανασταλεί εν μέρη. Και μάλιστα η κρίση του 90, ε, μας θυμίζει την κρίση του 90, τον πρώην Ιουκοσλαβικό πόλεμο. Εκεί ε, ε, η Κροατία, μια μικρή χώρα, περιέθαλψε 600.000 πρόσφυγες από την πρώην Ιουκοσλαβία και κυρίως από τη Βοσνία. Και ελάχιστοι από αυτούς πήγαν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν έλυσε το πρόβλημα της Βοσνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια εξωτερική δύναμη. Ίδια κατάσταση έχουμε και σήμερα. Η κάθε χώρα μένει ε, στο έλεος ε, και προσπαθεί να αντιμετωπίσει μόνη της ε, την κρίση όπως μπορεί. Όπως η κρίση στη Ιουκοσλαβία οδήγησε στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα τη Ευρωπαϊκής Άμυνας, ελπίζω η παρούσα κρίση να οδηγήσει σε καλύτερες κοινέ πολιτικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Χουντής η μέχρι σήμερα διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την ευρωπαϊκή ένωση συνιστά υπεκφυγή και υποκρισία. η ηγεσία της ευρωπαϊκής ένωσης κινείται κυρίως στην κατεύθυνση της καταστολής και λιγότερο στη λογική της αλληλεγγύης με αποτέλεσμα να συντηρούνται οι συνθήκες που έχουν μεταβάλει τη μεσόγειο το αιγαίο σε πλωτά νεκροταφεία. η ευρωπαϊκή ένωση έχει περιοριστεί σε ένα άχαρο ρόλο να παζαρεύει ανθρώπινες ζωές αρνούμενη να αντιμετωπίσει ένα εκρηκτικό πρόβλημα με ανθρωπιστικέ διαστάσει. Κύριε Αντιπρόεδρε, χρειάζονται γενναίε αποφάσει για τη δημιουργία ανοιχτών δομών φιλοξενία και τη διεκδίκηση του δικαιώματο των προσφύγων να φτάνουν με ασφάλεια στου ευρωπαϊκού προορισμού. Η επιμονή στην εφαρμογή του ξεπερασμένου συστήματο του Δουβλίνου θα οδηγήσει στην παραπέρα εγκλωβισμό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, κυρίω στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι η κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και η αντικατάστασή του από ένα σύμφωνο αλληλεγγύη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών η δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων κατάθεση αιτήσεων μετανάστευση πληστείων των περιοχών πολεμικών συγκρούσεων και η αλλαγή του χαρακτήρα τη frontex. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, συνάδελφοι. Μάλιστα. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχουν διαπράξει μεγάλα ασφάλματα. Αλλά τώρα αυτό δεν μας βοηθάει. Πρέπει να λύσουμε σήμερα ένα πρόβλημα το οποίο δεν αναγνωρίσαμε πολύ από εμάς και για λόγους που έχει να κάνει με τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και το δικαίωμα ασύλου. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες δικαίωμα και δεν υπάρχουν σύνορα ούτε προς τα πάνω. Όλοι έχουμε τη σύμβαση της Γενέβης και τις περισσότερες περιπτώσεις και στα συντάγματά μας. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι που έρχονται να έχουν μια ανθρώπινη συμπεριφορά με γρήγορες διαδικασίες και όχι μόνο σωστή αντιμετώπιση αλλά και όσοι δεν είναι πρόσφυγες θα πρέπει γρήγορα να επαναπροωθούνται. Ε, και εδώ είπαμε και για τη δική μου χώρα που καθυστερούμε. Θα πρέπει και εκεί να βάλουμε κάποια τάξη. Αλλά ποιο είναι το αποφασιστικό. Να ασχοληθούμε με τα αίτια αυτής της κρίσης. Οι πολίτες δεν πρόκειται να το δεχτούν εάν ε, αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα και να λύσουμε και τα προβλήματα και με το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συνομιλίες εχθές με την Τουρκία. Ωραία. Θα πρέπει να πούμε ε, ε, αν δεν, θα ε, τερματιστούν αυτοί οι πόλεμοι δια σε Ιράκ και σε Συρία δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα ε, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι βομβαρδίζουν σε τέσσε, τέσσερις χώρες βομβαρδίζουν. Ο καθένας βομβαρδίζει και κάποιον άλλον όμως στη Συρία. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Ε, χρειάζεται μια συνολική πολιτική, μια νέα πολιτική για την Αφρική, μια νέα εμπορική πολιτική για την προστασία και, ε, του κλίματος. Γιατί έχουμε και κλιματικούς πρόσφυγες. Όλα αυτά ε, να τα προτείνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες συνολικά. Αλλιώς θα μας στείλουν όλους σπίτια μας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε αυτή τη συνολική προσέγγιση και να το εξηγήσουμε και στους πολίτες. Θα παρακαλούσα και πάλι να σέβεστε το χρόνο σας, διότι τώρα προβλέπονται οι ψηφοφορίες τη μία παρατέταρτο, αλλά με όλους αυτούς τους ομιλητές που έχουμε, αν δεν σέβεστε το χρόνο αγόρευσης, θα πάμε μετά τη μία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε το χρόνο που σας έχει δοθεί. Ο κύριος Μωράης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω το τίτλο της σημερινής συζήτησης, αντίθετα με κάποιους συναδέλφους και χαιρετίζω τα όσα είπε η κυρία Μακάβεν. Είναι η πρώτη φορά που η εξωτερική διάσταση και αυτό το οποίο συζητάμε εδώ στα πλαίσια της πολιτικής συζήτησης έχουν ε, ειδωθεί από κοινού και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός πως ο κύριος Τίμερμαντς αναφέρθηκε στην ανάγκη της επίγουσας φύσης του θέματος γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά ε, τα μίντια απασχολούνται με την σύγκρουση στην Συρία μπαίνουμε στο χειμώνα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σημαίνει περισσότεροι θάνατοι στην Μεσόγειο ε, στις χερσαίες οδούς και αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην κρίση. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο θα πρέπει να αναθεωρήσει τους, να εξετάσει μάλλον τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και να θεωρήσει το θέμα αυτό επίγον. Θα ήθελα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερ και να του πω πως θα πρέπει να δούμε όχι μόνο ε, την, ε, το μηχανισμό επανεγκατάστασης αλλά και το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε πιο σωστά με το θέμα του οδικού χάρτη για την δημιουργία αυτών των hot spot έτσι ώστε να ε, είμαστε σίγουροι πως θα ακολουθήσουμε τις ε, σωστότερες λύσεις έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ορατά και για τους πολίτες στην Ευρώπη. Φορέντσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω τα εξή. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται λίγες μέρες μετά την τραγωδία ε, στη Λαμπεντούσα είναι κάποιες σφαγές για τις οποίες δεν μιλάει κανείς ποτέ. Τι οδήγησε στα εκατοπτώματα στο Λιβικό Πέλαγος. Ε, πόσα χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν τελικέ ακτές. Η μοναδική επίγουσα ανάγκη που έχουμε είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές αποφεύγοντας σφαγές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Η Ευρώπη δεν κάνει ό,τι πρέπει για να σώσει τις 120.000 ζωές που έχουν χαθεί παρηγορητικά και υποκριτικά είναι τα όσα λέμε όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των πολιτικών ε, προσφύγων, των οικονομικών μεταναστών, των μεταναστών προβλημάτων ε, από το κλίμα. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα καινούριο τείχος ε, μέσω του Δοβλίνου και πιστεύω πως θα πρέπει να καταστρέψουμε αυτό το τείχος και να δώσουμε οδούς για να περνάνε αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη θα πρέπει να τη χάνουν αξιοπρεπού μεταχείριση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τι ανθρωπιστικέ μα προσπάθειε για να στηρίξουμε την Ιορδανία, αλλά και τη Σερβία και τη Μακεδονία. Θα πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα κονδύλια στην υπατερμοστία το, για του πρόσφυγε και το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα και να στηρίξουμε και περιφερειακά προγράμματα. Δεν αρκεί να υποσχόμαστε κονδύλια. Θα πρέπει να εκταμιεύονται ταχύτατα τα κονδύλια και με συνοπτικέ διαδικασίε. Ούτε η ανθρωπιστική βοήθεια των hot ή επιτόπου στα κέντρα υποδοχής είναι αρκετή. Πήγα στη Λαπεντούζα και οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Μεσόγειο είναι αποτελεσματικές χάρη ε, στην συνεργασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τις τελικές αρχές και τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε ζωές και να καταπολεμήσουμε τους διακινητές που αλλάζουν όμως τον τρόπο ε, δραστηριότητάς τους. Θα πρέπει και εμείς ε, να εγκληματιστούμε στις αλλαγές. Επίσης ε, να δούμε το, νότιο δρόμο από την Τουρκία, την Αίγυπτο προς την Νότια Ιταλία και την Ελλάδα. Δυστυχώ, ε, τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν του κανόνε που ισχύουν και είναι σωστοί. Οπότε ε, η επανεκατάσταση είναι η καλύτερη σωστή λύση και από ένα σύστημα οικειοθελούς θα πρέπει να περάσουμε ένα σύστημα υποχρεωτική υποχρεωτικής Επίση ε, θα πρέπει η καταγραφή και η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων να γίνεται στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι στοιχείο θεμελιώδου σημασία για να λειτουργήσει το σύστημα Schengen. Ο αντιπρόεδρο σα όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχει νόημα να απευθύνουμε εκκλήσεις προς ξενόφοβους. Ε, κύριε Τίμερμανς, ε, το Συμβούλιο δέχτηκε την επιχειρηματολογία ε, υπέρ της υποδοχής των προσφύγων. Θα πρέπει όμως να πάμε πιο μακριά. Η ευθύνη και καθήκον μας είναι να δώσουμε σάρκα και οστά στα αποτελέσματα του Συμβουλίου, να τα μετατρέψουμε σε σωστές πρακτικές και πολιτικές και να έχουμε και μια πραγματική δύναμη πολιτικής προστασίας ε, στην Ευρώπη με συντονισμό των εθνικών ε, μονάδων. Γιατί η υποδοχή δεν σημαίνει απλώς ότι ανοίγουμε τα σύνορα ε, και παίρνουμε ανθρώπου. Χρειαζόμαστε και συνοριοφύλακες, θωριοφυλακή για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συνόρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Δύναμη Πολιτικής Προστασίας και Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Απαραίτητα μέτρα στα οποία θα πρέπει να εγκύψουν ταχύτατα το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλει τάχιστα πρόταση. Κυρία Γκαμπριέλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να χαιρετήσω την αύξηση των κονδυλίων για τη Frontex και για την Europol, αλλά θα ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή ε, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των οργανισμών και των κρατών μελών ε, και επίση και την εκπαίδευση των νέων προσφύγων γιατί είναι σημαντικό για να ενταχθούν. Επίση χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη για τα θύματα για να μπορέσουν πραγματικά να βγάλουν ε, ε, πέρα. Και επίσης οι γειτονικέ όμορες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, να τους υποδέχονται 130.000 ε, φοιτητές λέει Σαουδική Αραβία ε, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δίνουν κάποιους αριθμούς αλλά ε, πέρα από όλα αυτά εμείς τι κάνουμε για να απαντήσουμε με έναν τρόπο συνεκτικό σε αυτή την κρίση θα πρέπει να χαιρετήσουμε τις καταπληκτικές προσπάθειες που καταβάλουν Λίβανος και η Ορδανία είναι τεράστιες οι δυσκολίες αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κρατούν γερά αυτές οι χώρες. Ε, θα πρέπει να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας για να καταλάβουμε πώς μπορούν σήμερα αυτές οι χώρες να είναι νησίδες σταθερότητας ε, στην Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται να αυξήσουμε το παγκόσμιο πρόγραμμα για τα τρόφιμα θα πρέπει τα hot spot να εφαρμοστούν με το σωστό τρόπο για να μπορούμε να εντοπίζουμε, να δακτυλοσκοπούμε και να κατανέμουμε με αξιοπρέπεια τους πρόσφυγες. Τουρκία, εταίρος κλειδί. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση μας στη μάχη κατά της λαθρέας και παράνομης μετανάτευσης, κατά των διακινητών και ε, για να προσφέρουμε βοήθεια στους πρόσφυγες. Τι βοήθεια θα πρέπει να είναι ανθρωπιστική, συντονίζοντας με την υπατιαρμοστία, με τη UNICEF και με τις ευρωπαϊκές ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις τα διαφορετικά ταμεία της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να χτιστούν οι απαραίτητες υποδομές και τεχνικά με εμπειρογνώμονες από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Σε νομικό επίπεδο ενισχύονται τις διαδικασίες ασύλου για τον ε, έλεγχο των συνόρων, Κοινωνικοί για να μπορούν να ενταχθούν κοινωνικά οι μετανάστες ε, με πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Μία διάσκεψη δωρητών και τέλος η Ελλάδα χρειάζεται ειδική βοήθεια και διαφοροποιημένη βοήθεια για την περίπτωσή της. Κύριος Κοέγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια έκτακτη ανάγκη ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως είπε και ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος Τίμερμαν. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά τίποτα δεν έγινε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία, υπέβαλε καλέ προτάσει, αλλά στο Συμβούλιο ο Υπουργό Σμιτ, ε, όταν αποφάσισε τελικά, ελάχιστα μίλησε γι' αυτό και ελάχιστα έκανε. Απαιτείται από το Συμβούλιο να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε κρίση συνόρων, αλλά προσφυγική κρίση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ανάγκη βελτίωση τη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να δούμε πού θα δώσουμε τα κονδύλια εκεί, προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν αρκούν μόνο τα χρήματα. Επίσης, ε, ε, δεν είναι οι πρόσφυγες αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα Σέγγεν, αλλά τα κράτη-μέλη που δεν το εφαρμόζουν. Και ούτε 120.000 πρόσφυγες ε, θα, και η υποδοχή τους θα μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει το ρόλο της θεματοφύλακα της συνθήκης και να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων του Σέγγεν και της νομοθεσίας του ασύλου. Επίσης, να συνεργαστούμε με γειτονικέ χώρες, με τις χώρες της πρώτης γραμμής, να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου Πρέπει να συνεργαστούμε. Ουδέποτε δεν ήταν τόσο επιτακτική ανάγκη τη συνεργασία όπω σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Σβέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι διάβασα με έκπληξη αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ότι λέει ότι θα σταματήσει πλέον να δέχεται πρόσφυγες η Γερμανία και θα αρχίσει να τους απορρίπτει. Και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Σε χώρες δηλαδή που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ποιες χώρες υπάρχουν χώρες φιλικές προς τους πρόσφυγες και αναφέρθηκαν η Σλοβενία και η Κροατία. Μα δεν έχουν δυνατότητες απορρόφησης, είναι μικρές χώρες αν έχει την πρόθεση η Γερμανία να αποκρούσει ε, πάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες και να τους στείλει Σλοβενία και Κροατία, δεν γίνεται εμείς να τους υποδεχτούμε και να τους φιλοξενήσουμε. Παρακαλώ να τα ξανασκεφτούμε αυτά τα πράγματα και η Γερμανία να έχει και μια αντίστοιχη μεταναστευτική πολιτική όπως αρμόζει. Τώρα περνάμε στο Catch the Eye. Η κυρία Σοϊντρόβα. pane Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο. Πρέπει να σας πω ότι μετά από τα λόγια θα πρέπει να περάσουμε στη δράση. Στην ε, Τσεχία δεν υπάρχουν αντιδράσεις στα όσα ακούστηκαν στο Συμβούλιο. Θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη και θα πρέπει να προσφέρουμε με αλληλέγγυο τρόπο ανθρωπιστική βοήθεια. Η Τσεχία έχει ορίσει, έχει διαθέσει μάλλον, έχει περιχαρακώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει με το θέμα των μεταναστών ε, και κυρίως με το θέμα των προσφύγων από τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες. Γιατί για παράδειγμα δεν έχει ε, συμπεριληφθεί ε, η Αίγυπτος. Γιατί? γιατί στην Αίγυπτο παρόλα αυτά έχουμε χιλιάδες πρόσφυγες, οπότε εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε και ελπίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει μια γρήγορη απόκριση έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους αυτούς ανθρώπους με μια σύντομη έγκριση του προπολογισμού για να ε, βοηθήσουμε στις, ε, ε στους καταβλισμούς. Ευχαριστώ η ανθρωπιστική κρίση χρειάζεται αντιμετώπιση, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Θα με ακούτε, το μικρόφωνο λειτουργεί. Έχουμε λοιπόν μια ανθρωπιστική κρίση που συνδέεται με τη μετανάστευση και τα μέτρα που προβλέπονται είναι ένα καλό βήμα αλλά δεν αρκεί. Υπάρχει ένα θέμα που δεν συζητάμε. Οι ε, ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα παιδιά, ε, τα παιδιά συνολικά είναι 100.000 και έχουν αυξηθεί και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, έχουν διαπλασιαστεί, διαπλασιαστεί από πέρσι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προστατεύονται όπως άλλωστε ορίζει και το δικαστήριο θα πρέπει στην ε, επανεγκατάσταση ε, να ε, επιμείνουμε προς τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους που βρίσκονται στην επικράτειά τους ανεξαρτήτως χώρας πρώτης εισόδου ή χώρα στην οποία υποβλήθηκε έτσι ασύλου. Επίση, η οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για του ασυνόδευτου ανηλίκους για να μην πέφτουν στα χέρια και στα νύχια εγκληματικών οργανώσεων, όχι ε, μόνο πριν φτάσουν στην Ένωση, αλλά και όταν βρίσκονται στην επικράτειά του. Ο κύριος Μαριάς. Η κατάσταση των χιλιάδων προσφύγων που κατακλείζουν την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη είναι απελπιστική. Τα προσφυγικά κύματα αυξάνονται και η δυστυχία θα μεγαλώνει όσο θα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία, όσο θα ανέχεται και θα αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ίσις να συνεχίζει το εγκληματικό του έργο. Η ανθρωπιστική κρίση όμως δεν πλήττει μόνο τους πρόσφυγες, πλήττει και τον ελληνικό λαό που έχοντας φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια και την Τρόικα δεν μπορεί πλέον να φιλοξενήσει άλλους πρόσφυγες. Η Τρόικα όμως συνεχίζει να εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό με το τρίτο μνημόνιο και ενώ έπρεπε να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός που δέχεται τα τεράστια προσφυγικά κύματα ενώ έπρεπε να καταργηθεί το μνημόνιο και να διαγραφεί το επονίδιστο χρέος εσείς κύριοι της τρόικας και της κομισιόν συνεχίζετε να πιέζετε μαζί με το eurogroup την ελλάδα να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο και μετατρέπετε την ελλάδα σε κοινωνικό νεκροταφείο. αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο κύριος Γιακόφτσης. Σίγουρα στην τελευταία, στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής έγινε σημαντική πρόοδος. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της προσφυγικής κρίσης ε, υιοθέτησε μια πολύ καλή θέση και υπέβαλε προτάσεις για να λύσει αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Βέβαια, ε, δεν μπορούμε παρά να ομολογήσουμε την ε, έλλειψη ετοιμότητα και το πόσο απροετοίμαστοι είμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι δυστυχώ ε, και με τεράστια διαφορά ετοιμότητα μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να, ε, να λάβει πολύ πιο ηγετική ρόλο στον κόσμο στην επίλυση αυτής της κατάστασης και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ε, η Σερβία, η η Μακεδονία, έκαναν πολύ περισσότερα από ό,τι μερικές ε, ε, χώρες μέλη και πολύ περισσότερα από ό,τι... Το ίδιο πολύ περισσότερα από τις χώρες μέλη έπρεξαν η Ορδανία, ο Λίβανος. αν δεν κάνουμε κάτι πιο δραστικά θα συνεχιστεί η κατάσταση. Ο κ. Η, αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφυγοποίησης και της μετανάστευσης είναι ανεπαρκής και είναι και άνηση σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη. Από τα 2,4 δισεκατομμύρια που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα σχετικά προγράμματα τις τελευταίες εβδομάδες, για την Ελλάδα εγκρίθηκαν 470 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό, αν και φαίνεται μεγάλο σε απόλυτο αριθμό, είναι μόλις το 1 πέμπτο του συνόλου, τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα από την αρχή του 2015 έως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχει δεχθεί περίπου 310.000 καταγεγραμμένους ανθρώπους σε σύνολο περίπου 430.000 για ολόκληρη την Ένωση. Δηλαδή η Ελλάδα υποδέχεται τα 2 τρίτα του συνόλου των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και από την άλλη μεριά παίρνει μόνο το 1 πέμπτο των κονδυλίων για το σκοπό αυτό. Πρέπει να αλλάξουν αυτές οι αναλογίες. Κύριε Σκάρβερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η κρίση η μεταναστευτική είναι το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα των τελευταίων εποχών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εξέβρεση της καλύτερης λύσης και για τους πολίτες της Ένωσης και τους ίδιους μετανάστες. Ποιο είναι το πρόβλημα. Η Σαουδική Αραβία ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, μας είπε κάτι ίξης ε, αφήξης. Δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Γενέβης και δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η κρίση. Περιμένουν και στη Συρία και στο Λίβανο άλλοι ένα με 1,5 εκατομμύριο που ήδη ε, προωθούνται προς την Ευρώπη. Τα κράτη του κόλπου θα πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις για να δοθούν λύσεις ε, μόνιμες. Όλα τα κράτη-μέλη ε, των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να κυρώσουν τη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόμπερ Μάια γίνεται λόγο για ένα, με 1,5 εκατομμύριο μετανάστες φέτος για τη Γερμανία. Και το τσουνάμι αυτό το προσφυγικό δεν έχει τέλος. Ούτε διαφαίνεται. Και αυτό δεν είναι αξιοπερίοδο γιατί από Γιούνκερ μέχρι Τίμερμανς και Μέρκελ μέχρι Φάιμαν όχι μόνο τους προσκαλούν αλλά τους ε, υποδέχονται θριαμβευτικά. Δισεκατομμύρια θα κοστίσουν αυτά τα ανοιχτά σύνορα γιατί αυτό σημαίνει κόστος για αυτούς που έρχονται και λιγότερα χρήματα για τους φτωχούς της Ευρώπης και τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη που παραμένουν. Θα πέσει λοιπόν το βιωτικό επίπεδο και το κοινωνικό και στις πλούσιες χώρες της Ευρώπης και αυτό θα ε, θέσει ένα αμφιβόλο και θα απειλήσει την κοινωνική ειρήνη. Προσοχή λοιπόν. Έχουμε και ε, προοδό και επέλαση της Ισλαμοποίησης και του Ισλαμικού κράτους. Είναι εγκληματική αυτή η αμέλεια και η, η άγνοια. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκούσαμε διάφορα πράγματα για την Ουγγρική κυβέρνηση και για τον Βίκτορ Όρμπαν. Μπορεί να σας αρέσει, να μην σας αρέσει και Όρμπαν και η κυβέρνηση, αλλά αυτό που έχουμε είναι μάζες ε, λαθρομεταναστών ή λαθροπροσφύγων και ο κύριος Όρμπαν και η Ουγγρική κυβέρνηση εκπροσωπούν εκατομμύρια Ούγγρων πολιτών αλλά και εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη χώρα μας και επίσης θέλουμε να προσπίσουμε και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Μήπως να το θυμούνται αυτό και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοι ότι υπάρχει κάτι που παλιά το λέγαμε δημοκρατία διότι οι θύνοντες ε, δεν αποφάσιζαν στο παρελθόν με βάση τα όσα έλεγε μια μικρή ελίτ ή τα μέσα αλλά φογκραζόταν τον κόσμο και το λαό παλαιότερα. Και μιλούσαμε και για ελευθερία της γνώμης κάποτε. Και οι φίλοι μας στη Δύση όλα αυτά τα θεωρούν φυσιολογικά να κατακλυζόμαστε από αυτά τα τσουνάμι των προσφύγων ο πρόεδρο, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τίμερμανς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια σχόλια για να αντιδράσω στα όσα υπόθηκαν. Θέλω καταρχήν να είμαι σαφής. Έχουμε μια τεράστια κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε και είναι σαφέστατο πως η Ευρώπη δεν, δεν είναι σε θέση να δεχτεί όλους τους πρόσφυγες του κόσμου. Αυτό πρέπει να το πούμε απερίφραστα. Θα ήθελα... Συγγνώμη, ηρεμήστε, ηρεμήστε λίγο. Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Ο κανονισμός προβλέπει πέντε ε, παρεμβάσεις στη διαδικασία Catch the Eye. Έδωσα ένα πλέον ομάδα, αλλά παραπάνω δεν γινόταν. Ήδη είμαστε, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, γι' αυτό δεν μπόρεσα να δώσω το λόγο σε όλους όσους ζήτησαν τον κόσμο Catch the Eye. Παρακαλώ, μην διακόψουμε πάλι τον κύριο Τίμερμανς. Δεύτερον. Ε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν θα σας δώσω το λόγο, αλλά το λόγο έχει ο κύριο Τίμερμαν, ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, λοιπόν, η ανθρωπιστική κατάσταση σημαίνει πως θα πρέπει να δράσουμε σε όλα τα επίπεδα. Τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των κρατών μελών αλλά και εκτός αυτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί ανέλαβε ηγετική δράση στο θέμα αυτό και για τη στεναρή στήριξη στις θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Εάν κάνουμε αυτά τα οποία συμφωνήσουμε και τα κάνουμε ταχύτατα, ναι, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και θα δείξουμε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, πώς θα τα καταφέρουμε, πώς η Ευρωπαϊκή Εύρωση μπορεί. Τρίτον, για κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Εάν δεν επιθυμείτε να βοηθήσετε τους πρόσφυγες ή εάν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα παρά μόνο να τους αποθείτε στα σύνορα, πείτε το. Και μην προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε παριστάνοντας πως αυτοί που φτάνουν στην Ευρώπη δεν είναι πρόσφυγες. Είναι ψέμα. Τουλάχιστον έχετε το θάρρος της γνώμης σας βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Μην λέτε πω οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πρόσφυγες. Το 80% των ανθρώπων που φτάνουν σήμερα στην Ελλάδα μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Of course. η κρίση των προσφύγων φέρνει και προβλήματα. Κανεί δεν το αρνείται και τα προβλήματα αυτά θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να βελτιώσουμε τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να είμαστε πολύ ταχύτεροι με τη δαστηλοσκόπηση, με την ταυτοποίηση των ατόμων και με γρήγορο τρόπο να επιλέγονται αυτοί που έχουν δικαίωμα ε, στην χορήγηση ασύλου και όσοι δεν έχουν να επιστρέφονται ε, ε, στη χώρα από την οποία προήλθαν. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδε. Αλλά το να φωνάζει κανεί από τον πάγκο και να λέει αυτοί οι κακοί άνθρωποι θα πρέπει να εξαφανιστούν από τα ραντάρ δεν θα προσφέρει καμία λύση στο πρόβλημα. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έγιναν πολλά σχόλια για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μία επιστολή διοικητική στις Ουγγρικές Αρχές για να μας ξεκαθαρίσουν τι γίνεται με ένα, μια σειρά ζητημάτων για τα όσα κάνουν με τον έλεγχο των συνόρων και με την επεξεργασία των ζητημάτων ασύλου. Περιμένουμε και μετά θα προχωρήσουμε σε διάλογο με τις Ουγγρικές Αρχές επί τη βάση της απάντησης που θα μας στείλουν. Ο κύριος Νικολάς Σμίτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πρόσφυγες πολέμου δεν επιλέγουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Δεν έχουν απλούστατα άλλη επιλογή. Εμείς βοηθούμε λοιπόν στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας τους εκτοπισμένους όσο γίνεται ε, πιο κοντά στις αιστείες τους. Και όταν υποχρεώνται να διαφύγουν προς τρίτες χώρες γειτονικές, εκεί θα πρέπει κατά προτεραιότητα να τους βοηθήσουμε. Ακόμα και η ανθρωπιστική βοήθεια πάντα δεν επαρκεί. Θα πρέπει να αποφύγουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό οι άνθρωποι αυτοί απεγνωσμένοι να μπουν σε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη που έχει κοστίσει ήδη πάρα πολλές ζωές. Εγώ θα ήθελα να αναρωτηθούμε. Ρωτήστε έναν οικογενειάρχη. Ε, ε, όταν ρωτήθηκε ένας γιατί ε, το σε αυτό. Και απάντησε, γιατί τα παιδιά μου επί δύο χρόνια δεν έχουν πάει σχολείο. Εγώ ρωτώ όλους εκείνους που αρνούνται την πραγματικότητα, όπως μόλις είπε ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς θα περιμένατε δύο χρόνια για να μπείτε σε αυτό το ταξίδι. Αυτή η ανθρωπιστική κρίση, όντως, όπως πολύ υπογραμμίσατε, απευθύνεται σε στις αρχές και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες είμαστε βαθύτατα προσιλωμένοι. Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού, ε, αναζητώντας απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι στεναρή, αποτελεσματική, συνολική και στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρώπη είναι σε θέση, είναι να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και θα το πράξει μόνο εφόσον είναι αλληλέγγυη. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώνεται και περνάμε στις ψηφοφορίες. Uh, Συνάδελφοι, θα περάσουμε στις ψηφοφορίες, αλλά προηγουμένως ε, ο κύριος Μαμαζαγιάς ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, Ζήτησα το λόγο όντω, γιατί το, βράδυ ε, Σαββάτου προς Κυριακής ε, στο διαμέρισμα Alp Maritim στην Νότιο Γαλλία είχαμε τρομερές καταιγίδες και πλημμύρες, κατακλυσμό ουσιαστικά. Είχαμε ε, τεράστιες ηλικές ζημιές, 20 θανάτους, ε, μερικούς αγνοωμένους και θα ήθελα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη αλληλεγγύης ε, προς τη Γαλλία. Δεδομένου όμως ότι θα έρθει αύριο ο πρόεδρος Ολάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα το Κοινοβούλιο να εκδηλώσουν προς την Γαλλία και τις χώρες που έχουν πληγεί από τα καιρικά αυτά φαινόμενα αύριο τη συμπαράστασή τους, την συμπάθεια και τη φιλία τους προς τους συναδέλφους, προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μας επισημάνατε αυτή την τραγωδία στη Γαλλία και σας ε, διαβεβαιώ ότι αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα το θέσει όπως πρέπει. Κύριε Έριξον, διαδικαστικό. Υπάρχει πρόβλημα με το κατάλογο ψηφοφορίας, ε, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση Γκάιερ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου από ό,τι ξέρω την ανέλαβε την έκθεση στην Επιτροπή Προπολογισμών ε, εισηγητής ε, που κατάγεται από την ίδια εκλογική περιφέρεια στην οποία εδρεύει η επιχείρηση που ζητά την, για την οποία γίνεται κινητοποίηση. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Θα έλεγα λοιπόν να αφαιρεθεί το σημείο από την ημερήσια διάταξη ή τουλάχιστον ο Πρόεδρος να συζητήσει αυτό το θέμα στην Αρμόδια Επιτροπή ή με τους πρόεδρους επιτροπών ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Γιατί νομίζω ότι έχουμε μια κατάφορη περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Δεν νομίζω ότι θέλει να απαντήσει ο κύριος Γκάιερ στο σχόλιο, οπότε ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Α, βλέπω ακόμη ένα διαδικαστικό όμως. Έχετε διαδικαστικό ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο απολύτω με την ψηφοφορία. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Και είχαμε πει ότι όταν έχουμε περίπτωση μιας χώρας που μας αφορά, δεν θα... σαν, να... σαν λέμε ότι όταν έχουμε περίπτωση μιας χώρας που μας αφορά, δεν δικαιούμαστε να λαμβάνουμε μέρος στην ψηφοφορία. Θα πρέπει να έχουμε επαφή των βουλευτών με τους πολίτες και σας διαβεβαιώ ότι δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα με πτώση στη διαδικασία αυτή και τίποτα παράνομο. Ωραία, ας περάσουμε στην πρώτη